πρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για την κατάσταση στην Μολδαβία. Παραμένουμε λοιπόν στην ίδια περιοχή της Ευρώπης κατά το μάλλον ήτον. Τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο Στυλιανίδη σχετικά με την Μολδόβα, την Μολδαβία. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ολομέλεια το θέμα της χώρας αυτής από την επικύρωση εδώ και ένα χρόνο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Πολλά γεγονότα έλαβαν χώρα από τη συζήτηση του περασμένου έτους, μεταξύ των οποίων το Νοέμβριο 2013 ε, ε, εκλογών και είχαμε δύο κυβερνήσεις που είχαν μικρή διάρκεια ζωής. Όλοι σας έχετε παρακολουθήσει από τότε την, ε, την κατάσταση στη χώρα αυτή, κυρίως όσον αφορά ε, την, ε, την, το θέμα των τραπεζών που, και το, θέμα, το πρόβλημα που ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Και βεβαίως, με συγχωρείτε, περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια, που 12% του ΑΕΠ της χώρας. και βεβαίως είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στην αρχή του Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη ε, συνάθρηση στο Τσιτσινάου. Ενώ αυτό το σκάνδαλο, ε, το τραπεζικό, ήταν στο επίκεντρο των διαδηλώσεων, ο λαός εξέφρασε ευρύτερα τη δυσφορία του, ζητώντας βιώσιμη κυβέρνηση και ζητώντας την καταπολέμηση της διαφθοράς με τρόπο αποφασιστικό παρά μια μείωση της έντασης ε, κυρίως με αναμονή των πολιτικών εξελίξεων ε, αυτές οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση του Προέδρου επίσης ε, την εκδίωξη του Γενικού ε, Εισαγγελέα και των αρχών κατά της διαφθοράς και ζητούν ε, την προετοιμασία ενός δημοψηφίσματος για να υπάρξει άμεση εκλογή του Πρόεδρου. Οι πρόσφατες εξελίξεις, κυρίως η σύλληψη του πρώην Πρωθυπουργού Φίλαν στις 15 Οκτωβρίου και η ε, μετέπειτα διάλυση της κυβέρνησης ε, με ψήφο δυσπιστίας δείχνουν δραματικά την ε, μεγάλη ρήξη που υπάρχει ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, τα οποία και στις κυβερνήσεις που ήταν κυβερνήσεις συνασπισμού. εφόσον δεν είναι ρόλος μας να αναμειγνιόμαστε στις εσωτερικές διαδικασίες μιας ε, χώρας κυριέρχης, πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις της Μολδαβίας ε, να αφήσουν κατά μέρο τα ενδιαφέροντά τους προς όφελος της χώρας, εναπόκειται σε αυτές να κάνουν τις πολιτικές επιλογές που θα λαμβάνουν υπόψη την ευημερία των πολιτών, να βοηθήσουν στον εξυγχρονισμό ε, της χώρας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί και είναι έτοιμη να υποστηρίξει θα συνεχίσουμε να ζητούμε ένα διάλογο μεταξύ των κομμάτων, ούτως ώστε να βρεθούν βιώσιμες λύσεις στην κυβερνητική κρίση και βεβαίως ούτως ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν πιεστικές ανάγκες. Ελπίζουμε ότι μια νέα κυβέρνηση θα δώσει άμεση προτεραιότητα στην εφαρμογή και υλοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων και ότι ε, πρακτικές διαφθοράς ε, και η διαπλοκή ε, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας και έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η κοινωνία της Μολδαβίας περιμένει να αντιμετωπιστούν σοβαρά αυτές οι προκλήσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα της της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Σύνδεσης στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου του περασμένου Σεπτεμβρίου και επίσης είχαμε ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ΑΦΕΤΑ και του ε, Προέδρου του Κοινοβουλίου Γκαντού στην αρχή της περασμένης εβδομάδας θα πρέπει να θυμίσουμε στους εταίρους μας της Μολδαβίας ότι η υποστήριξή μας δίδεται υπό όρους βάσει της υλοποίηση πραγματικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα πρέπει να συμβάλλουν όχι μόνο ε, στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, αλλά ε, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια χώρα πιο στιβαρή, πιο ανθεκτική και ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Κάθε νέα κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση του να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό του σκανδάλου με, αμερόληπτη, με αμερόληπτες έρευνες και ολοκληρωμένες ούτως ώστε να ανακτηθούν τα κονδύλια, τα κεφάλαια. Η κοινωνία της Μολδαβίας περιμένει κάθε νέα κυβέρνηση να λάβει μέτρα σοβαρά κατά της διαφθοράς και ζητάει την μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα και τη δημόσια διοίκηση. Η Μολδαβία βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση και χρηματοπιστωτική και θα χρειαστεί τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπληρώσει ορισμένους όρους σχετικά με τα τι ενεργειακά τιμολόγια, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα ταυτόχρονα ε, την, ε, και την ε, διαχείριση της Εθνικής Τράπεζας αυτή είναι προϋποθέσεις προαπαιτούμενα απαραίτητα ε, για να υπάρξει υποστήριξη του προϋπολογισμού από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε ε, την φιλόδοξη ατζέντα σύνδεσης που έχουμε. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται τα, στα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, στις σχέσεις του πολιτικού συστήματος με την κοινωνία. Είναι σοβαρό το θέμα, γι' αυτό θα πρέπει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσουμε να υλοποιηθούν τα προαπαιτούμενα που ανέφερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα περνάμε στους αγωγητές των πολιτικών ομάδων. Πρώτα-πρώτα, εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο πρόεδρος Έλμαρ Μπρόκ, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο, κύριε Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Αγαπητοί επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω, κύριε επίτροπε, ότι με την παρούσα περιγραφή που δώσατε για τα θέματα της Μολδαβίας έχετε δίκιο. Πρέπει να μεριμνήσουμε τα τρία ευρωπαϊκά κόμματα που κέρδισαν στι, τις εκλογές με μικρή διαφορά αλλά παρόλα αυτά κέρδισαν δεν ήταν όμως σε θέση από την άλλη πλευρά να ε, οικοδομήσουν την, ε, ε, την εμπιστοσύνη των πολιτών και δεν ήταν σε θέση τους στόχους του εξυγχρονισμού της χώρας για το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεν ήταν σε θέση να σημειώσουν κάποια σημαντική πρόοδο. Από την άλλη τώρα πλευρά, υπάρχουν πολλοί σε αυτά τα κόμματα που έχουν την προθυμία πρέπει να πω να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και από πλευρά κοινοβουλευτικών εκπροσώπων μπορούμε να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί ώστε να υπάρξει μια φιλευρωπαϊκή κυβέρνηση επιτέλους που θα αναλάβει τα ενία της χώρας διότι οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν ολέθρια και γι' αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι, πολιτικοί, οι πολιτικές οικογένειες αυτού του σώματος θα πρέπει σε σχέση και με τα κόμματα να βρουν το θάρρος να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν τους όρους αυτής της συνεργασίας ώστε η Μολδαβία να μπορέσει να λάβει τις αποφάσεις για λογαριασμό της, ποια κυβέρνηση θα δημιουργήσει, όμως πρέπει να υπάρχει μια προσφορά συνεργασίας από πλευράς μας. Και γι' αυτό τον λόγο θα υπάρχει η ελπίδα. Η ευθύνη και η υπευθυνότητα όλων στη Μολδαβία θα τους κάνει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε αυτό θα είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν είναι χρόνος να αναζητήσει κανείς το προσωπικό του κέρδος και ιδιοτέλεια, ούτε για κομματικά παιχνίδια. Είναι μιας χρονική στιγμή για δέσμευση, ανάληψη δεσμεύσεων προ όφελο ε, του μολδαβικού του λαού, του λαού τη Μολδαβία. Και ελπίζω ότι οι διαβουλεύσει και οι συζητήσει που θα διεξαχθούν αυτέ τι ημέρε θα οδηγήσουν σε τέτοιε αποφάσει. Και αυτό δεν θα αποτύχει λόγω των εξαρτήσεων και πολιτικών ε, ε, ιδιαιτεροτήτων, να στις αποκαλέσω έτσι, και θα έχουμε μια θετική έκβαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, των Σοσιαλδημοκρατών, Κριστέα παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπο, πριν από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναντήθηκε για να επικυρώσει τη Συμφωνία Σύνδεση. Με αυτόν τον τρόπο, ε, ο οίκο μα αναγνωρίζει τι προσπάθειε μεταρρύθμιση και τι ε, φιλοδοξίε των μολδαβικών αρχών. Σημειώθηκε πρόοδο και η επικύρωση ήταν ένα σημαντικό ε, μήνυμα αναγνώρισης. Η Μολδαβία ήταν ε, από τους πρωτοπόρους της Ανατολικής Γειτονίας ε, και μια επιτυχής ιστορία τότε. Σήμερα συναντώμαστε για να μιλήσουμε για την Μολδαβία, αλλά όχι για να γιορτάσουμε την πρώτη επέτειο από την επικύρωση. Για να το πω, μα δεν υπάρχει κανένας λόγος να γιορτάσουμε τίποτα. Ε, τους τελευταίους 12 μήνες ε, συνάντησα τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Ο πέμπτος ετοιμάζεται να αναλάβει. Ο συμπρόεδρος τη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργός ε, συνελήφθη με κατηγορίες διαφθοράς. Ε, ένα σκάνδαλο τραπεζικό με τις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες ε, οδήγησαν στην εξαφάνιση ενός δισεκατομμυρίου περίπου το 50% του ΑΕΠ της Μολδαβίας. Και τώρα που η χώρα και ο λαός χρειάζονται ε, αποφασιστική δράση και όραμα από την πολιτική τάξη, περισσότερο παραποτέ τα κόμματα δεν είναι σε θέση να προτείνουν ούτε καν ένα, μια νέα κυβέρνηση, ένα νέο πρωθυπουργό. Η κατάσταση είναι σοβαρή, τόσο σοβαρή που ο πειρασμός είναι να θυμώσουμε το Κισινάου, γιατί μας απογοητεύει. το θαύμα έπαψε να είναι θαύμα. Αλλά θα πρέπει να αντισταθούμε για χάρη των πολιτών της Μολδαβίας. Αξίζουν κάτι περισσότερο, αξίζουν τη δέσμευσή μας, την ενθάρρυνσή μας και θα είμαστε στο πλευρό τους περισσότερο από ποτέ. Η πολιτική τάξη της Μολδαβίας απλώς απογοήτευσε τους πολίτες και ανησυχούμε τα μάλα. Η πολιτική διαδικασία ε, είναι απρόβλεπτη, η πολιτική κατάσταση είναι σε μόνιμη κατάσταση αστάθειας ε, σε χρόνια φάση ε, κρίσης. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Οι ανάγκες του πληθυσμού δεν αντιμετωπίζονται, οι μεταρρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και οι πολίτες ε, πληρώνουν τα σπασμένα. Η Μολδαβία χρειάζεται κάποιους υπεύθυνου πολιτικούς ηγέτες. Χρειάζεται διαφανείς θεσμούς. Για να το πω απλά, η Μολδαβία χρειάζεται μια πολιτική τάξη που είναι σε θέση να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μια νέα ε, κυβέρνηση η οποία ε, θα μεταφράζει την ε, Συμφωνία Σύνδεσης και θα εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει κράτος δικαίου, ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαιοσύνη, καταπολέμηση με σοβαρότητα της διαφθοράς, διερεύνηση του τραπεζικού σκανδάλου και να δικαστούν οι υπεύθυνοι. Είναι τελευταία ευκαιρία για την απερχόμενη κυβέρνηση συνασπισμού. Πέρασε η προθεσμία και δεν υπάρχει εναλλακτική παρά μόνο να συνεχιστούν οι σημερινές μεταρρυθμίσεις. Εμείς και οι πολίτες Μολδαβίας βλέπουν ότι χρειάζεται να δράσουν οι υπεύθυνοι και θα πρέπει να το καταλάβουν και οι πολιτικοί ηγέτες της Μολδαβίας. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέλντερ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόσφατα είχαμε επισκεφθεί την Μολδαβία και ως ε, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όταν επισκέπτομαι χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνία, συνεργασίας και εταιρική σχέσης με τέτοιου είδους αποστολές όταν πηγαίνω πρέπει να πω ότι σπάνια έζησα μια τέτοια κατάσταση όπως αυτήν στο Κίσιναο, πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Ρώτησα τον πρέσβη, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για αυτή την κατάσταση και η απάντησή του ήταν όχι. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα. Και ταυτόχρονα αυτή η πολιτική χρεοκοπία πρέπει να πω ότι ουσιαστικά έχει επιπτώσεις και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάντα αναφερόταν ότι είμαστε φίλοι εμείς. Πρόκειται για σημαντική απώλεια εμπιστοσύνης λοιπόν έναντι της Ευρώπης και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να δούμε με ποιους συναλλασσόμεθα και με ποιους διαβουλευόμεθα σε σχέση με την Μολδαβία. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Στην χώρα μου υπάρχουν εδώ και δεκαετίες χριστιανικά ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα που ενδιαφέρονται και μεριμνούν για τους ε, πτωχούς ε, και πιο αδύναμους. Και δόξα τω Θεώ μπορούν με τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες να διατηρήσουν, να διασφαλίσουν το κύρος μας και μπορούμε γι' αυτό να είμαστε περήφανοι για τη Μολδαβία για αυτές τις προσπάθειες. Στη συνέχεια ο κύριος Αστρεβίτσιος παρακαλώ. Mr. Chairman, Mr. Commissioner. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο, όταν μιλούσα για την Μολδαβία, και ήμουνα εισηγητής, θυμάμαι ότι είχα πει ότι είναι πρωτεργάτης η Μολδαβία. Ε, ηγέτης της χώρας της Ανατολικής ε, Γειτονίας. Ήταν η πρώτη η οποία απολάμβανε ε, καθεστώς ε, χωρίς θεωρήσεις. Ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και Σύνδεσης με μας που άρχισε να λειτουργεί και να δίνει αποτελέσματα. Η Μολδαβία είχε όλα τα πολιτικά εργαλεία, τις τα έδωσε όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τονώσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μολδαβία. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά. Όλο και περισσότερο. Άνευ προηγουμένο αυτό το τραπεζικό σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σοβαρή έρευνα μέχρι στιγμής και πλήρης. Τα στοιχεία διαφθοράς σε όλους τους πολιτικούς ε, χώρους, σε όλα τα πολιτικά στρώματα, ε, μαζί με την ε, διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διάθεση για διερεύνηση. Τα πράγματα έχουν βαλτώσει. Οι, αλλάζουν οι κυβερνήσεις με την ταχύτητα που αλλάζουν οι εποχές του χρόνου. Σε μια τέτοια κατάσταση είναι φυσικό ο κόσμος να κατεβαίνει στους δρόμους και να παραμένει για μήνες. Το θέμα είναι πότε αυτή η ένταση θα οδηγεί σε έκρηξη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά από προτεργάτης η Μολδαβία έγινε σύμβολο χάους, πολιτικού χάους. Κάνω έκκληση σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τις ελίτ της Μολδαβίας να ξυπνήσουν. Ήγηκε η ώρα. Ξυπνήστε και δείξτε ότι έχετε ευθύνη πολιτική απέναντι στη χώρα σας και στο λαό σας. Ο λαός σας που αξίζει να ζήσει στην Ευρώπη και να απολαμβάνει τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος ο κύριος Σόλτς εξ ονόματος της ομάδας της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσα σε 7 χρόνια τέσσερις εκλογές ε, αλληλοδιάδοχες κυβερνήσεις και ατέλειωτες ε, αντιπαραθέσεις πολιτικών ηγετών και διαρκώς ε, διαφθορά. Αυτό λοιπόν πραγματικά πιέζει τους αναλυτές να βρουν μια εξήγηση. Και βλέπουμε ότι ο πρώην ιδιαίτερος ε, μαθητής, ο καλύτερος μαθητής έγινε θύμα των διεφθαρμένων ολιγαρχών. Να τονίσω ένα πράγμα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αν δεν είχε συμβεί αυτό δεν θα το είχε προσέξει ιδιαίτερα κανείς. Ωστόσο όμως η πολιτική αποτυχία δείχνει πόσο δεινή είναι η θέση αυτής της χώρας. Παρόλες τις εκλογές, λόγω της διαφθοράς, βρίσκεται σε διαρκή εξάρτηση από εξωτερική βοήθεια αυτή η χώρα πρέπει να δούμε ότι είναι διαρκώς εκλογές οι οποίες διεξάγονται και δεν μπορεί να λυθεί το θέμα της πολιτικής εξουσίας. Είναι ιδιαίτερα δαπανηρή αυτή η διαδικασία και η δικαστική εξουσία διαρκώς παραβιάζει τις αρχές όσον αφορά για παράδειγμα την αντιπολίτευση και τους ε, διαδηλώνοντες και διαμαρτυρόμενους κατά της ε, κατάστασης αυτής. Και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο περιορίζει τις ε, ελευθερίες του κράτους δικαίου. Και βλέπουμε εδώ ότι οι ε, μεταρρυθμίσεις ε, χωλένουν και βλέπουμε μια τάξη η οποία ναι μεν λέει ότι θέλει και πρόκειται να προπορεθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως συμπεριφέρεται όπως οι ολιγάρχες. Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπονομευθεί λόγω συσχετισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διεφθαρμένους πρέπει να επιμείνουμε να τηρηθούν οι αρχές της συμφωνίας. Αυτό, αναμένει, αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της Γεωργίας. Um, on behalf uh, Greens, uh, Ευχαριστώ εξ των Πρασίνων η κυρία Έντι Οτάλα. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται, ε, υπάρχει εδώ ε, στην ε, Μολδαβία υπήρξε μια σφιγμομέτρηση πάρα πολύ σοβαρή. Μόνο 39% αυτών που απέντησαν είναι θετική υπέρ της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ περίπου 43% ε, είναι υπέρ της προσχώρησης στην Ευρωασιατική Συμμαχία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης όπου ε, το κοινό έχει αρχίσει να ε, κουράζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται σαν συγκάλυψη πολυβρώμικων πολιτικών. Και σήμερα οι δύο ευρωπαϊκές οικογένειες, το ΕΛΚΑ και οι ΣΟΙΤΕΣ έχουν αναγνωρίσει ότι έχουν μια ευθύνη και χρησιμοποιούν τις επαφές τους για να εξηγήσουν ότι αυτό που γίνεται τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί δεν θα πρέπει να υπερισχύσει η ατιμορρασία σε αυτό το ε, απίστευτο τραπεζικό σκάνδαλο. 15% του ΑΕΠ αυτής της φτωχής χώρας ε, έχει χρησιμοποιηθεί ε, και έχει πάει σε χέρια ιδιωτικά. Οι ένοχοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα πρέπει να μπορεί να πληρεί το λειτουργήμά της. Με συγχωρείτε κύριε Θερτσεβίτσιος, Ρουνάνσκι. Ε, σας παρακαλώ ε, να πάτε να συζητήσετε εκτός της αίθουσας. Κόρβιν και παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη Γεωργία χωρίς να μιλήσουμε για την την χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή του Ρωσικού στρατού. Και βλέπουμε ότι έχουμε και τις, ε, ε, το πρόβλημα το οποίο ανακύπτει. Τι θα γίνει σε σχέση με αυτή την περιοχή οι υπήκοοι της Μολδαβίας που δεν επιθυμούν να υπάρχει αυτή η κατάσταση ιδιαίτερα δεδομένη της μεγάλης διαφθοράς δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπήκοοι της Μολδαβίας διότι γνωρίζουν ότι είναι προφανές ότι όπου υπάρχει λέει δημοκρατία υπάρχει και διαφθορά όπου λοιπόν υπάρχει δημοκρατία υπάρχει διαφθορά και έχουμε δύο διαφορετικές κοινωνίες εκείνους στη Μολδαβία που δεν γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ας τους αφήσουμε λοιπόν στη μοίρα τους. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε και μπορούμε να προχωρήσουμε με τον κύριο Πρέντα παρακαλώ. Έχετε τον λόγο κύριε Πρέντα. Ε, mai mulți colegi s-au referit la faptul Ευχαριστώ. Πρέπει να πω και να αναφερθώ ότι μέσα σε ένα έτος η δημοκρατία της Μολδαβίας από πρωτοπόρος προπομπός της ε, ανατολικής γειτονίας έγινε ουραγός ε, Κάποιο, ο οποίο δηλαδή δεν είναι πλέον προβλέψιμος και επικρατεί χάο στη Μολδαβία. Πώς καταλήξαμε σε αυτήν την κατάσταση. Πιστεύω τρεις σημαντικοί παράγοντες υπάρχουν που επηρεάζουν και αλλάζουν την κατάσταση στη Μολδαβία. Πρώτα, η Ρωσία ίδια η επιρροή της ε, Ρωσίας ε, που ασκείται στην κοινή γνώμη είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Δεύτερον, οι ολιγάρχες οι οποίοι ελέγχουν, ελέγχουν τα πολιτικά κόμματα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι κατά το παρελθόν. Τρίτον, η διαφθορά. Η διαφθορά που αποδυνάμωσε τα θεσμικά όργανα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι κατά το παρελθόν πάλι, πριν δηλαδή από τις εκλογές του Νοεμβρίου μπορούμε να δούμε την αποτυχία, έκδηλη, εξόφθαλμη αποτυχία του φιλευρωπαϊκού συνασπισμού που κέρδισε τις εκλογές και που καταβλήθηκε η προσπάθεια ναι με να λειτουργήσουν οι οργανισμοί και οι θεσμοί όμως δεν τα κατάφεραν και ενισχύθηκε, ενδυναμώθηκε η πολιτική κρίση από αυτό. Έχουμε ευθύνε λοιπόν και ο Έλμαρ Μπρόκ ανέφερε, αναφέρθηκε στις πολιτικές οικογένειες να υπομισθούν τις ευθύνε που έχουν Ωστόσο να μην το ζητάμε αυτό από τους κομμουνιστές. Η κομμουνιστική οικογένεια στο Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να μπει στο περιθώριο και όλοι οι φίλοι της Ρωσίας στο Κοινοβούλιο οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το ολέθριο σενάριο για τη Μολδαβία θα έπρεπε να ζητηθεί να παραμείνουν εκτός να μείνουν στο περιθώριο, να μην αναμειγνύονται. Να ρωτήσουμε τι πρέπει να γίνει με το Κίσιναο, να διαμεσολαβήσουμε για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού συνασπισμού, μιας νέας πολιτικής συμμαχίας να προσφέρουμε με τις προσπάθειές μας και με την αναθεωρημένη πολιτική γειτονίας μια προοπτική για τη Μολδαβία και τις άλλες γειτονικές χώρες. Πρέπει να εμπλακούμε και να, να συνδιαλλαγούμε με τους μετριοπαθείς με εναλλακτική πορεία σε σχέση με αυτό που επιθυμούν οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές για τη Μολδαβία. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευρωβουλευτά Πρέντα. Νίνα Γκυλ παρακαλώ θα λάβει τον λόγο. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Οι Μολδαβοί πολίτες έχουν εντοπίσει τις προτεραιότητες τους. Όταν ε, κατέβηκαν στον δρόμο τον περασμένο μήνα για να πέσει η κυβέρνηση. Η διαφορά είναι το πρόβλημά τους. Είναι προς το συμφέρον τους να το αντιμετωπίσουν ε, και προς το συμφέρον μας, γιατί είναι κατά της ε, ασφάλειάς μας, γιατί η Μολδαβία είναι σημαντικός κόμβος για το λαθρεμπόριο όπλων. Όχι μόνο Καλάσνικοφ, οι εγκληματίες ε, προσπαθούν να πουλήσουν κλαμμένα, ε, κλεμμένα, κλεμμένα πυρηνικό υλικό στο Ισλαμικό κράτος και σε άλλους τζιχαντιστές. Ε, μία απόπειρα απαιτεύχει από το FBI, αλλά άλλες μπορούν να πετύχουν. η αστυνομία της Μολδαβίας που ερευνά Ε, αυτή την, ε, αυτό το έγκλημα, ε, σταμάτησε το ρευνά γιατί την εμπόδισε η κυβέρνηση. Γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να υπάρξει μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και αυτό να γίνει απόλυτη προτεραιότητα. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς που θέλουν να, να ελέγξουν τους θεσμούς για προσωπικό όφελος να, να τους κάνουμε εταίρους μας ακόμα και αν είναι υπέρ των ευρωπαϊκών πολιτικών. Φυσικά, μην ξεχνάμε τη Ρωσία, η οποία παίζει το κλασικό τη παιχνίδι. Και παίζει τα, χρησιμοποιεί του ανθρώπου ω πιόνια. Αλλά δεν πρέπει ε, να παίξουμε το παιχνίδι των ε, ανθρώπων αυτών που δεν ε, θέλουν να λειτουργήσουν σωστά οι θεσμοί. Θα πρέπει να πούμε, εντάξει, προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις και τότε εμείς σας βοηθάμε. Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει όμως ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι προς, το προς ίδιον όφελος και δεν θα πρέπει να μπει στον πειρασμό να στρέψει την πλάτη της στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ αυτών που το παίζουν ε, σύμμαχοί της. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρσκι. Παράλληλα. Σας ζητώ, κυρίες και κύριοι, Να μην φέρνετε εδώ τα παλτά σα. Μπορείτε να τα αφήνετε έξω. Υπάρχει χώρος. E, Πρέπει να σεβόμαστε το χώρο τη Ολομέλειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Κάσκι, σα ευχαριστώ. Μια πολιτική κρίση βλέπουμε ότι είναι αυτή. Η κυβέρνηση απεπέμφθη και εδώ και μήνες έχουμε εντονότατες διαμαρτυρίες επειδή έχουν απογοητευτεί οι πολίτες από την κυβέρνηση. Και όλα αυτά δεδομένων των τεράστιων σκανδάλων διαφθοράς ε, που όπως γνωρίζουμε συνυπολογίζονται σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάπως από, ε, ε, απετέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης. Ιδιαίτερα η μεταρρύθμιση του διοικητικού σκέλους και της δικαιοσύνης και όλες οι μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πρόσφατα είχαμε και τον πρόεδρο της ε, Βουλής της Μολδαβίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τεκμηρίωσε αυτά τα γεγονότα. Υποστηρίζουμε φυσικά τη Μολδαβία προς την, σε σχέση με την ανατολική γειτονία και την πορεία τη, Ωστόσο πρέπει να καταστήσουμε σαφέ ότι υπήρξε ένα ορόσημο μέσω της συμφωνίας σύνδεσης. Ωστόσο η χώρα τώρα προσανατολίζεται προς άλλες αγορές, ε, ιδιαίτερα προς την Ρωσία. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση στο Κίσιναο θα συνεχίσει την καταπολέμηση, τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και θα εισακούσει τους πολίτες και ευχόμαστε στους ε, μολδαβούς εταίρους μας κάθε επιτυχία. Εμείς ως Πολωνοί γνωρίζουμε ότι οι στόχοι μπορεί να μην είναι εύκολοι να επιτευχθούν λόγω της πολιτικής πίεσης και έντασης και λόγω της πίεσης και έντασης που δημιουργεί η Ρωσία και μέσω της Απχαζίας ε, ε, και της υπερνηστερίας γίνεται η προσπάθεια να υπονομευθεί η χώρα. Είναι γνωστή αυτή η πολιτική πολιτική. Ευχαριστώ. Ε, στη συνέχεια ο κύριος Μαστάλκα παρακαλώ. E, e, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ ταραχώδης η κατάσταση στη χώρα αυτή και οι σχέσεις με τους γείτονες πάντα ήταν προβληματικές στην ιστορία της Μολδαβίας συν πολιτική διαφθορά και η ιδιωτικοποίηση που συνέβη κλιμάκωσε τα προβλήματα. Είναι βασικά γεωργική αυτή η χώρα. Παρά το γεγονός αυτός, αυτό, το μόνο που έλειπε ήταν μια συμφωνία για την ε, ανάπτυξη. Η Μολδαβία δεν θέλησε ποτέ να γίνει τμήμα της Ρουμανίας οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ε, επιθυμούν την ε, προσέγγιση της ε, με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη δεν έχει παίξει το πολιτικό της ρόλο για να εξαλείψει την διαφθορά στη χώρα αυτή. Ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα με τη γυναίκα του Προέδρου, την κυρία Πετρένκο. Ευχαριστώ. Σόλτες. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πέρασε ένας χρόνος από την υπογραφή της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ ΕΕ και Μολδαβίας για το εμπόριο και την ε, σύνδεση και τις δυνατότητες που θα διανοιγόντουσαν προλιένοντας το έδαφος ε, για τη Μολδαβία ώστε να υπάρχει ανταλλαγή εμπορευμάτων και ε, εργαζομένων. Πέρασε και ένας χρόνος από τότε που η αντιπροσωπεία μας πήγε στην Μολδαβία κατά τη διάρκεια της εποχής των φιλευρωπαϊκών δυνάμεων Ωστόσο όμως ε, απολέσει η εμπιστοσύνη του πληθυσμού σε αυτό το συνασπισμό και δεν υποστηρίζει πλέον την φιλευρωπαϊκή πορεία ε, ο πληθυσμός μια και αισθάνθηκε ότι προδόθηκε σε σχέση με τις προσδοκίες του αλλά έχουν αναφερθεί τα προβλήματα σε σχέση με την ελευθερία των μέσων του τύπου σε σχέση με την κατάσταση των τραπεζών του κράτους δικαίου και αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα είναι ε, το ότι βρίσκονται στους δρόμους και διαμαρτύρονται και η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος Μίχαελ Γκάλερ έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Γκάλερ. Σε σχέση με τη Μολδαβία, πολλά στοιχεία του λόγου μου για τη Γεωργία δυστυχώ μπορούν να επαναληφθούν. Η Μολδαβία είναι σημαντική για μα, ο σημαντικό γείτονά μα. Οι πολίτε τη Μολδαβία είναι σημαντικοί για μα ω Ευρωπαίοι, επειδή βρίσκονται σε εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζονται και θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα. Θέλουμε να ενταχθούν οι πολίτε τη Μολδαβία στο δικό μα οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, διότι έτσι αυξάνεται η ζώνη της γειτονίας μας. Η εμπλοκή μας ε, σε σχέση με τη Μολδαβία δεν είναι άνεφόρων και προϋποθέσεων. Αναμένουμε σεβασμό του κράτους δικαίου, αναμένουμε σεβασμό για τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία καθαρή και έντιμη πολιτική. Αυτές τις προσδοκίες έχουν επίσης οι πολίτες της Μολδαβίας οι Μολδαβοί τον ε, εξυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις ε, ε, τους, τις υποστήριξαν. Αναμένουν εξυγίανση ενώ οι ολιγάρχες παλεύουν να διατηρήσουν την εξουσία τους. Κυρίως οι πολίτες αναμένουν μια διακρύβωση των εγκλημάτων. Πού βρίσκονται τα δισεκατομμύρια που εκλάπησαν από τις τράπεζες. Θα ελπίζαμε οι μυστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών να διέθεταν στοιχεία στην Μολδαβία ώστε να μπορέσει να εντοπιστεί πού βρίσκεται αυτό το χρήμα χρήμα και να επιστραφεί στη Μολδαβία. Χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση η Μολδαβία. Χρειάζεται ένα ισχυρό ανεξάρτητο γενικό εισαγγελέα και καταπολέμηση τη διαφθορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει αυστηρού όρου και προποθέσει. Μια εξειδικευμένη συνθήκη θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να, προβλε... να ε, δρομολογηθούν οι μεταρρυθμίσει και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Η υποστήριξή μα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση αυτών των όρων και προποθέσεων. Η οι πολίτες της Μολδαβίας ε, θέλουν να αλλάξει η κατάσταση. Δεν επιτρέπεται να απολέσει και άλλους πολίτες η Μολδαβία. Δεν θέλουμε να απολέσουμε τους Μολδαβούς. Ε, δεν θέλουμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Και γι' αυτό θα ήθελα από πλευρά του ΕΡΚ να ασκηθεί η επιρροή μας ε, στα κόμματα που έχουμε επαφή μαζί τους, ώστε να ασκηθεί η επιρροή μας υπέρ αυτής της ημερήσιας διάταξης του θεματολογίου που καταρτήσαμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ. και στη συνέχεια τον Κλαουδιάν Φρουζουλίκα παρακαλώ. Ε, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μιλήσω στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, την ρουμανική γλώσσα. Ε, οι παραδόσεις, ο ε, πολιτισμός, η γλώσσα ε, τα ανθρώπινη δεσμή, η γεωγραφία, η δημοκρατία της Μολδαβίας είναι μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και όχι της γεωγραφικής περιοχής της Ευρωασιατικής. Η δημοκρατία της Μολδαβίας έχει προβλήματα, αλλά δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτρέψει ε, την δημοκρατία της Μολδαβίας σε μια περιοχή φόβου, αστάθειας με την Ουκρανία. Όπως ξέρετε, η δημοκρατία της Μολδαβίας Μολδαβίας έχει μια παγωμένη διένεξη από το 1991. Η Ουκρανία πιο πρόσφατα έχει το θέμα της Κρυμαίας και τώρα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία της Μολδαβίας για να έχει μια βιώσιμη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να ωφεληθούν από την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούν να δουν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο, με τον ευρωπαϊκό κόσμο ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν εκεί συμφέροντα που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη δημοκρατία της Μολδαβίας. Πρέπει να, τους, να τα καταπολεμήσουμε, να υποστηρίξουμε βιώσιμη κυβέρνηση στο Κίτσινάου, να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών που είναι φιλοευρωπαϊκή. Η δημοκρατία της Μολδαβίας θα πρέπει να προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και η Ρουμανία. Το μέλλον της είναι η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πέτερ Έριξον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Μολδαβία πρέπει να αναφέρουμε είναι μια όμορφη χώρα με απίστευτο δυναμικό ωστόσο όμως και με σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτύχαμε στο να αντιμετωπίσουμε στις, ε, την ευρύτατη αυτή διαφθορά στη Μολδαβία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας ε, καταδιώκει. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σκάνδαλο των τραπεζών να φωτιστεί, να διαφωτιστεί, να γίνει η διακρύβωση εκείνη που θα οδηγήσει, θα προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι 12, του, ε, ποσοστό 12% του ΑΕΠ εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Αυτό είναι απόλυτα παράδεκτο. Και εδώ τονίζεται το ότι η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινωνία έχει ε, απολεστεί. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα δηλαδή. Πρέπει να είναι σαφές ότι θα προσφέρουμε οικονομική και νομική βοήθεια ώστε οι υπεύθυνοι να προσαρθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν και να δημιουργηθεί ένα λειτουργού σύστημα τραπεζικό για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο Ευρωβουλευτής κύριος Πλένκοβιτς. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που ο λαός της Μολδαβίας εξέφρασε την φιλοδοξία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα και έλλειψη μεταρρυθμίσεως και ε, έχασαν πολλά πράγματα. Υποστηρίξαμε την Μολδαβία με τρόπο πολιτικό και οικονομικό, αλλά η κατάσταση είναι απαράδεκτη επειδή η πολιτική ελίτ έφερε τη χώρα ε, στο χείλος του γκρεμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης που της Μολδαβίας που είναι τώρα η η φτωχότερη χώρα και έχουμε εκεί ολιγάρχες σε όλα τα ε, κυβερνητικά όργανα. Η καταπολέμηση της διαφοράς, η, μετάβαση οικονομική, η δημοκρατία είναι προτεραιότητες που υποστηρίζονται από, από την πλειονότητα του λαού. Θα πρέπει να κάνουμε έκκληση στην πολιτική ελίτ και θα ήθελα να επικροτήσω τα όσα είπε ο κύριος Μπρόκ και ο κύριος Οστρεβίτσι ότι όλες οι δυνάμεις υπέρ των μεταρρυθμίσεων πρέπει να οργανωθούν και να στρέψουν την προσοχή τους στη Συμφωνία σύνδεση. Μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα βοήθεια στην Μολδαβία όπως έχουμε και με την Ουκρανία και να παρατείνουμε την θητεία που θα είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα για την Μολδαβία. Η κατάσταση στην υπερδνηστερία είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και θα πρέπει να επανέλθουν τα πράγματα σε ευρωπαϊκή τροχιά. Πλάνκοβιτς, ευχαριστώ και τώρα δίνω τον λόγο στον Σίκφριντ Μούρασάν Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Όποτε βρίσκομαι στη Μολδαβία, ο κόσμος μου με ρωτάει το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Η Μολδαβία υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει. Είναι καθήκον ως εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών να προσφέρουμε στη Μολδαβία μια ευρωπαϊκή προοπτική και στους πολίτες της ε, χώρας αυτής να τους δώσουμε ελπίδα, να τους δείξουμε ότι έχει ελπίδες. Εάν δεν τους δώσουμε προοπτική, θα τους δώσει προοπτική ο Πούτιν. Και δεν θα είναι καλή αυτή η προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ή για τη Μολδαβία. Η δημοκρατία της Μολδαβίας ε, υποφελείται από την Συμφωνία Σύνδεσης και από την προσέγγιση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα όμορη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι δικαιούχος ε, των περισσότερων κονδυλίων κατά κεφαλήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες της Μολδαβίας πόσο επωφελής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς και πόσο πιο επωφελές είναι το να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε την προπαγάνδα που τους λέει πηγαίνετε προς τη Ρωσία. Το 2014 όταν η Ρωσική Ομοσπονδία επέβαλε εμπάργκο σε μολδαβικά προϊόντα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε και τους επέτρεψε να εξάγουν περισσότερα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε ένα αξιοπρεπέ βιωτικό επίπεδο στου εξαγωγεί και στους ε, γεωργού. Πρέπει να τους πούμε ποιο είναι φίλος, ποιο είναι εχθρός. Πρέπει να τους πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια ανεξάρτητη και ισχυρή ε, Μολδαβία. Ευχαριστώ κύριε Μουρασάν. Και τώρα ο επόμενος ομιλητή, Κοσλόφσκα Ρασέγιουτ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, κυρίε και κύριοι, Περίπου πριν από ένα έτος ε, η Μολδαβία υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ. Ως πρώτη χώρα της ανατολικής γειτονίας η χώρα απέκτησε πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και διευκολύνσεις διαβατηρίων, θεωρήσεων διαβατηρίων. Ήταν ικανοποιητική αυτή η οδός. Τους επόμενους μήνες είδαμε ότι ένας πολιτικός σεισμός ε, συνέβη στην ε, Μολδαβία διαδηλώσεις στο Κισινάο για τις κλοπές και τη διαφθορά κατά τη ελίτ όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις προς όφελος των ολιγαρχών. Αυτό οδήγησε στην πτώση της φιλευρωπαϊκής κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση έπρεπε λοιπόν να αποπεμφθεί και έτσι η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια φθήνουσα πορεία και σε σχέση με την κατάσταση ήταν μια πολύ σοβαρή κρίση η οποία εξεράγει. Και αυτό την χώρα αυτή την ε, κατέστησε ευάλωτη έναντι αλλοδαπής ανάμειξης και επιρροής ε, όπως της Ρωσίας. Αξίζει κάτι καλύτερο η Μολδαβία. Να είναι σε θέση δηλαδή να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης. Διότι μια λειτουργούσα δικαιοσύνη είναι αποφασιστική σημασία. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι υπάρχει η δικαιοσύνη και ότι οι εγκληματίες θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Και τίθεται το ερώτημα, τι μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τι μπορούμε συγκεκριμένα χειροπιαστά να προσφέρουμε ως υποστήριξη στη Μολδαβία για να βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη ρωσική προπαγάνδα που διαθέτει στοιχεία προς επηρεασμό των πολιτών. Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων η Μολδαβία. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, η Μολδαβία ήταν ε, επιτυχική, επιτυχής ε, ιστορία όταν εφάρμοσε την Συμφωνία Σύνδεσης ε, με απελευθέρωση. Αλλά οι ηγέτες της έκαναν πολλά λάθη. Η... Τα αίτια συνδέονται με το παρελθόν. Η έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας μεταξύ των πολιτικών ελίτ. Έχασαν την αξιοπιστία τους, χάσαν τα λεφτά από τις τράπεζες, χάσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών ένα χρόνο μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Δεν υπάρχει ενότητα ε, για να υπάρξει ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Οι πολιτικές ελίτ δεν έχουν πια τη δύναμη να ηγηθούν της χώρας. Αποφάσισαν τώρα να αναγγείλουν νέες εκλογές χωρίς να μπορούν να προβλέψουν τα αποτελέσματα. Εμεί είμαστε με τους Μολδαβού. αλλά χρειαζόμαστε επιχειρήματα για να προωθήσουμε την ένταξή τη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι καθήκον μα να του ε, υποστηρίξουμε προ τη μεταρρύθμιση. Ε, μέτρα κατά τη διαφθορά, να υπάρξει συμφωνία με το ΔΝΤ του για να συνεχίσουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής βοήθειας για τον, για τον ισορροπημένο προϋπολογισμό. Όπως είπε και ο Μπροκ, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους Μολδαβούς για να βρουν το σωστό δρόμο μόνοι του. Θα μπορούμε να περάσουμε, ψηφί... να μπορούμε να περάσουμε ψηφίσματα, αλλά είναι και η ώρα για μια νέα ηγεσία, μια ηγεσία εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Κύριε Μπόνη, ξεπεράσατε το χρόνο σας. Κατά 52%. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Στανισλάβ Πόλτσακ, πρώτος και καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, τονίσω το χάος, την πολιτική αστάθεια στην Μολδαβία επί του παρόντος και τι θα έπρεπε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τη Μολδαβία μετά τις βουλευτικές εκλογές το 2014 και την πτώση δύο κυβερνήσεων και μετά από τόσες κατηγορίες διαφθοράς και κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να έχουν μια εναλλακτική λύση οι Μολδαβοί. Ιδαλλιώς θα στραφούν, ξέρουμε που αλλού μπορούν να στραφούν. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγρότες στην Μολδαβία όπως προσπαθήσαμε να το πράξουμε πάρα πολλές φορές, αλλά και αυτό που θα πρέπει επίσης να κάνουμε πάνω απ' όλα είναι να τους προσφέρουμε κάποια προοπτική ε, στην επόμενη περίοδο και να τους δείξουμε ότι είμαστε στο πλευρό τους. Ευχαριστώ κύριε Πόλτσακ. Uh, κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Μολδαβία είναι έκρηθμη. Την ώρα που έχουν δημιουργηθεί τεράστια οικονομικά προβλήματα στη χώρα. Την ώρα που η διαφθορά ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω στο πολιτικό σύστημα. Την ώρα που πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν ως διαμαγείας από το τραπεζικό σύστημα και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό την ώρα που μένεται η πολιτική κρίση μετά την ανατροπή της κυβέρνησης υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος η μολδαβία να κυλήσει σε βίαιες εσωτερικές συγκρούσεις των δύο μεγάλων πολιτικών μπλοκ που κυριαρχούν στη χώρα από τη μια πλευρά εκείνων που επιθυμούν μια στενότερη σχέση με την ευρωπαϊκή ένωση μέσω της ανατολικής εταιρικής σχέσης και από την άλλη πλευρά όσων επιθυμούν να βλέπουν το μέλλον τους κοιτώντας ανατολικά η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να συμβάλλει στην εμπέδωση της δημοκρατίας στο χτύπημα της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου χωρίς όμως να επεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική κατάσταση και στις κομματικές αντιπαλότητες στη μολδαβία. μόνο έτσι μπορεί η ευρωπαϊκή ένωση πράγματι να συμβάλλει στην πολιτική ηρεμία στην περιοχή. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Τελευταίος ίδια γλώσσα, αλλά όχι ίδια χώρα. Εκ μέρους της Επιτροπής, ο Επίτροπος ε, κύριος Στυλιανίδης, Χρήστος Στυλιανίδης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, to thank you for... να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας, για την υποστήριξή σας και την αποφασιστικότητά σας. για το πολύ δύσκολο και επίμαχο θέμα που μαστίζει μια χώρα της γειτονία μας με πολλές επιπτώσεις. Η συζήτηση μας σήμερα επιβεβαιώνει ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες όλοι μας και ότι χρειαζόμαστε να υποστηρίξουμε τη Μολδαβία στην πορεία της για την πολιτική σύνδεση και οικονομική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις προσπάθειές της να δημιουργήσει μια δημοκρατική κοινωνία και να ξεπεράσει τα συμφέροντα των μεμονωμένων ατόμων. Προς το συμφέρον της χώρας όμως. Η κοινωνία της Μολδαβίας περιμένει από τους ηγέτες της να θέσουν τέρμα σε αυτή την ομοιρία του κράτους, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, να κάνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις και να ανακτήσουν τα κλεμμένα ποσά από τις τράπεζες. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τη Μολδαβία σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Μόνο όμως η πολιτική της Μολδαβίας μπορεί να υλοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Μαζί με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, τα προναφερθέντα είναι εκ των για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα της χώρας. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την αποφασιστικότητά σας στο πλευρό της Μολδαβίας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.